<laughs> Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte Platz. Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινούμε με την κοινή μας συνεδρίαση μαζί με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και φυσικά και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, γνωμοδότηση της ε, νομικής υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την συμβατότητα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά με το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο το οποίο έλκεται από τις συνθήκη της Λισαβόνας. Χαίρομαι λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι για την παρουσία σας και από τις δύο <clears throat> επιτροπές ώστε να μπορέσουμε από κοινού να συζητήσουμε για τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν πρέπει να το κάνουμε και κλεισμένο των θυρών αλλά δημόσια και να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας δημόσια. Η συμφωνία με τον Καναδά βρίσκεται στην τελευταία της φάση. Το Συμβούλιο θα επιληφθεί του θέματος αυτού την επόμενη εβδομάδα συζητήσαμε και εμείς στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και εάν εγκριθεί από το Συμβούλιο στις 18 Οκτωβρίου και η υπογραφή στις 27 Σεπτεμβρίου η συμφωνία, θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει σε βάθος αυτήν την ε, συμφωνία. Βέβαια πρέπει να ελεχθεί και ο χαρακτήρας αυτής της συμφωνίας και αυτό είναι και το αντικείμενο της ε, σημερινής μας ε, ε, συζήτησης και θα δώσω την, το λόγο στην νομική υπηρεσία, αλλά προηγουμένως στον συμπρόεδρό μου, κύριο Σφόμποτα. Σας ευχαριστώ κύριε Λάγκε και σας ευχαριστώ που συμφωνήσατε να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψε με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο ήταν και θέμα συζήτησης και στη δική μας Επιτροπή, τη Νομική Επιτροπή, σε διάφορες ευκαιρίες πρόσφατα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη νομική υπηρεσία για την θέλησή τους να συνεργαστεί μαζί μας. Το θέμα της ε, προστασίας των επενδυτών στη συμφωνία και η δημιουργία του δικαστηρίου για την επίλυση διαφορών, αυτά είναι τα θέματα για τα οποία είμαστε αρμόδιοι ως Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ως εκ τούτου προσβλέπουμε στη συζήτηση των θεμάτων αυτών και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ κοντά τι εξελίξει στο θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Και εγώ σα ευχαριστώ από τη δική μου πλευρά, λέει ο κύριο Λάγκε, για την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό από κοινού και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην νομική υπηρεσία ο κύριος Άντερ Νέγκαρτ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της αντίστοιχης μονάδος για 10 λεπτά μάξιμου για να μπορούμε να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε διότι Έχουμε περιορισμένο χρόνο. Στις 10 θα πρέπει να ψηφίσουμε. Κύριε Νέγκαρτ, για 10 λεπτά το πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ τους χρονικούς σας περιορισμούς. Η γνωμοδότηση αυτή λοιπόν αφορά τη συμβατότητα με τις συνθήκες, ιδιαίτερα με το ΣΕΤΑ. Δεν είναι δηλαδή μια γενική αξιολόγηση, κάτι το οποίο ο τίτλος θα μπορούσε να μας κάνει να σκεφτούμε. Κανονικά το ISDS είναι ένα δικαστήριο ad hoc που αποτελείται από πέντε διαιτητές νομικούς. Τώρα έχουμε αναπτύξει ένα νέο μέσο το οποίο περιλαμβάνει ένα μόνιμο δικαστήριο και περιλαμβάνει επίσης και έναν αριθμό νέων ρητρών ασφαλείας. Το θέμα είναι αν το σύστημα αυτό είναι συμβατό με τις συνθήκες και ιδιαίτερα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέγει ότι οι εθνικές συμφωνίες, οι διεθνείς συμφωνίες έχουν ε, προτεραιότητα σε σχέση με το δευτερογενές δίκαιο και το δικαστήριο ουσιαστικά το ευρωπαϊκό ε, έχει το μονοπόλιο σε σχέση με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Δεν είναι κάτι το νέο ότι οι διεθνείς συνθήκες αποδίδουν σε διάφορα είδη δικαστηρίων την δυνατότητα να αξιολογούν τις διεθνείς ή εθνικές συμφωνίες. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκφραστεί με την αποφάσεις του για την δυνατότητα αυτή. Ε, σημείο εκκίνησης είναι ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας ε, προβλέπουν την δυνατότητα προσφυγής σε δικαστικό σώμα, σε δικαστικό όργανο μάλλον, το οποίο προβλέπεται από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Όταν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες πληρούνται. Πιο συγκεκριμένα δεν θα πρέπει να υπάρχουν, ε, αν θέλετε, ε, επιπτώσεις αρνητικές στη νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να θίγονται οι αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων και δεν θα πρέπει να δεσμεύονται οι λειτουργίες των οργάνων αυτών σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου. Επιπλέον του θέματος της ερμηνείας του κοινοτικού δικαίου και μιλήσαμε ε, για το ε, μονοπόλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην αναγνώριση ευθυνών και σε εξοδικαστικό επίπεδο και εξετάσαμε επίσης αν υπάρχει εδώ δυνατότητα σύγκρουσης με, με ε, θέματα πρωτογενούς δικαίου και επίσης στήθεται και το θέμα της, ε, του καθορισμού των αρμοδιοτήτων και του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη σχετικά με την αυτονομία της ε, ενωσιακής νομικής τάξης. Σύμφωνα με την δικαστική διαδικασία Λούλιν και σύμφωνα με ε, συγκεκριμένο άρθρο της συνθήκης, αναγνωρίζεται ότι η αρμοδιότητα για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου δεν μπορεί να βαφεί σε οποιοδήποτε άλλο σώμα δικαστικό. Τώρα όμως η εφαρμογή ε, και οι συνθήκες εφαρμογής μιας διεθνούς συμφωνίας είναι κάτι το οποίο εφόσον συναποτελεί μαζί με άλλες ρυθμίσεις το κοινοτικό δίκαιο, ανήκει στις αρμοδιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ βλέπουμε ότι το δικαστήριο που δημιουργεί η ΣΕΤΑ είναι αρμόδιο για την ερμηνεία και την εφαρμογή των επιπέδων προστασίας των επενδυτών που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία και όχι ουδίποτε άλλου νομικού στοιχείου της Ευρωπαϊκής Νομικής Τάξης δεν επηρεάζει τη συμβατότητα του κοινοτικού δικαίου με οποιοδήποτε άλλο νομικό σύστημα, παρόλα αυτά στις αξιολογήσεις του το δικαστήριο αυτό μπορεί να λαμβάνει υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, αλλά μπορεί να το κάνει αυτό με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι δεσμευτικό σε σχέση με την ερμηνεία την οποία δίδει στο, ενωσιακό, σε εισαγωγικά δίκαιο δεν προβλέπεται δυνατότητα στη Συμφωνία ΣΕΤΑ της ε, ε, εκ των προτέρου διαβούλευσης ε, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι το ενωσιακό δίκαιο είναι το συγκεκριμένο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό και η γνωμοδότηση 2 κάθετος 13 σχετικά με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χάρτα στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το δικαστήριο είπε ότι ε, ο μηχανισμός αυτός απαιτεί πρώτερη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση όμως για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα ίδια θέματα, για τα ίδια νομικά θέματα, για τα οποία προβλέπονται ρυθμίσεις σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου. Coordination between those two aspects of it. So we had a set of rules which are fundamentally the same. Um, There was also, there's also the fact that the... Είναι σαφές επίσης ότι η Σύμβαση επιτρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν υψηλότερα επίπεδα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει αντικείμενο συντονισμού σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου. Υπήρξαν ε, κάποια προβλήματα σε σχέση με τις απαιτήσεις της σύμβασης να ελέγχονται ότι οι άλλες χώρες σέβονται τη σύμβαση. Και υπάρχει εδώ το θέμα της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Επιπλέον, το σύστημα το οποίο λειτουργεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις συμβουλευτικές επιτροπές ε, μπορεί να γίνει αντικείμενο εγγύησης από τη Σύμβαση, ε, κατά κάποιο τρόπο αγνοώντας το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο. Αυτά δεν προβλέπονται λοιπόν στα πλαίσια της ΣΕΤΑ. Νομίζουμε ότι η γνωμοδότηση 2 κάθετος 13 είναι, ένας, είναι μια ευκαιρία αναγνώρισης της συμβατότητας των ρυθμίσεων για το διατητικό δικαστήριο με το κοινοτικό δίκαιο. Σε σχέση τώρα με τις εξωτερικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεκδικήσεις στα πλαίσια του συστήματος προστασίας των επενδυτών της ΣΕΤΑ δεν βασίζονται ε, στις ε, επιπλέον αναλήψεις υποχρέωσης ευθυνών της Ένωσης ή στις εξωσυμβατικές ακριβώς ευθύνες και δεν φύγεται το πεδίο που είναι αποκλειστική, αν θέλετε, αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα μπορούσαν βέβαια να υπάρξουν ανησυχίες για το ότι αυτό το οποίο μπορεί να αποφασίσει το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι να υπάρξει οικονομική αποζημίωση για την παραβίαση των αρχών της προστασίας των επενδυτών. Τώρα, αν το οικονομικό βάρος είναι τόσο μεγάλο που επηρεάσει έμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σε οικονομικό επίπεδο, τότε θα μπορούσε να κηρυχθεί παράνομο. Όμως, βλέποντας το θέμα αυτό σε επίπεδο τυπικό, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο. Γιατί όχι μόνο προσθέτει, ε, δεν θα αποτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, λόγω ακριβώς του υψηλού οικονομικού κόστους που θα προκληθεί, να λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο. Σε μια ακραία περίπτωση, λοιπόν, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε μια παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Αλλά ε, η παραβίαση αυτή δεν θα παραβιάζει τις προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου, γιατί η ΣΕΤΑ περιλαμβάνει κάποιες ρήτρες προστασίας και αν κάτι δεν πάει καλά υπάρχει μηχανισμός διόρθωσης ε, της συγκεκριμένης παραβίασης του κοινοτικού δικαίου στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια αξιολόγηση ξεχωριστή σε σχέση με τις κρατικές βοήθειες, τις κρατικές επιδοτήσεις. Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια ε, λήψη υπόψη της έννοιας της οικονομικής βλάβης για μία από τις συμβαλόμενες πλευρές. Η απόφαση, σαν παράδειγμα, να διακοπεί μια επιδότηση ή να μην δοθεί μια επιδότηση δεν θα πρέπει να θεωρείται όμως παραβίαση. σε σχέση με τη ΣΕΤΑ. Ο καθορισμός τώρα των αρμοδιοτήτων προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει αν η Ένωση ή ένα κράτο μέλος πάρει μέρος σε μια δικαστική διαδικασία σε σχέση με μια διεκδίκηση. Έτσι λοιπόν οι συνταγματικές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα εδώ βλέπουμε ότι η προστασία των επενδυτών γενικότερα και στα πλαίσια της ΣΕΤΑ ε, καλά τώρα εντάξει να σταματήσω εντάξει. να προσθέσω ίσως κάτι να πω ότι ε, και το τελευταίο που πήγα να πω αλλά δεν είπα ρυθμίζεται από τη ΣΕΤΑ. Όλα ρυθμίζονται. Ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε ερωτήσεις ή δηλώσεις. Κάθε φορά ένα μέλος της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ και ένα μέλος της Επιτροπής Γιούρι. Από τη Γιούρι η κυρία Χαουτάλα παίρνει το λόγο πρώτη. Για δύο λεπτά το ανώτατο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει συζήτηση κατά πόσο πρέπει να έχουμε ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία μάλλον για όλα αυτά. Σίγουρα χρειαζόμαστε επενδύσεις και σίγουρα χρειαζόμαστε νομικό πλαίσιο. Αυτός όμως είναι ο σωστός τρόπος να ε, προχωρήσουμε. Είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το σύστημα επίλυσης επενδυτικών διαφορών έτσι όπως προβλέπετε. Δεν είμαι καθόλου πεπισμένη. Ο Γενικός Εισαγγελίας Κόκοτ ε, έχει γράψει γι' αυτό και θεωρεί ότι η διαιτησία μπορεί να είναι ε, προβληματική γιατί δεν είναι προαπαιτούμενο να εξαντληθούν τα νόμιμα εγχώρια ένδικα μέσα εκ των προτέρων πριν προσφύγει κανείς στη διαιτησία δεν μπορούν τα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά να ε, αποφανθούν και δεν δικαιούνται ε, όσοι ασχολούνται με την επίλυση των επενδυτικών διαφορών δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν την προκαταρκτική προδικαστική διαδικασία. Υπάρχει και η απόφαση 213, στην οποία αναφέρθηκε η νομική υπηρεσία. Αυτό καταρχάς λοιπόν είναι το πρώτο μου ερώτημα, η παρατήρηση. Δεύτερον, η προστασία των ξένων επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις στην εσωτερική αγορά. Εξ όσων κατάλαβα, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση εναντίον κρατών μελών σχετικά με το θέμα αυτό, ουσιαστικά δημιουργούνται διακρίσεις γιατί δίδεται προτεραιότητα στις ξένες επενδύσεις, στις επενδύσεις γενικότερα, εις βάρος των εσωτερικών επενδυτών της εγχώριας αγοράς. Ουσιαστικά ενθαρρύνουμε ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητά να αναδιοργανωθούν νομικά για να φαίνονται ως αν να είναι ξένες επενδύσεις. Ένας Σουηδός ή Φιλανδός επενδυτής επενδύσει, αν επενδύσει στην Ισπανική αγορά, μπορεί να κυκλοφορεί τα χρήματα μέσω μιας θηγατρικής του στην Σιγκαπούρη ή μέσω ενός οχήματος ειδικού σκοπού που να έχει συστήσει. Ε, υπ' αυτή την έννοια, για να μπορέσει να ε, έχει προστασία της επένδυσής του βάσει του συστήματος επενδυτικών δικαστηρίων και του ε, συστήματος επίλυσης επενδυτικών διαφορών. Θεωρώ ότι υπάρχει εκεί πεδίο για διακρίσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Κίρτον Τάρλιν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή της νομικής γνωμοδότησης. Παραμένουν τα ερωτηματικά για το κατά πόσο το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων και η ΣΥΤΑ συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχω συγκεκριμένο θα ερωτούσα και εγώ για τη μη διάκριση σε βάρος της εγχώριας της εσωτερικής αγοράς και για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, των οποίων ε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ανήκει π.χ. σε Καναδούς επενδυτές θα έχουν διαφορετικά δικαιώματα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά και αναρωτιέμαι και εγώ κατά πόσο εκεί ε, δίνεται λαβή για διακρίσεις, αλλά αφού τέθηκε αυτό το ερώτημα ήδη, θέλω να ρωτήσω τα εξής. Ποια είναι η γνώμη της νομικής υπηρεσίας για το ποιες συνέπειες θα έχει η σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας που να μην είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι θα συμβεί δηλαδή αν τελικά το Συμβούλιο συμφωνήσει στη ΣΥΤΑ και μετά υπάρχει προσφυγή στο Δικαστήριο του ευρωπαϊκό και το δικαστήριο αποφανθεί ότι όντως δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ότι μελλοντικά οι επενδυτικέ διαφορέ θα υπάρχει απόφαση ότι πρέπει να υπάρξει πληρωμή και το καθεξής. Και στη συνέχεια ρωτώ και το εξή. Μπορεί να υπάρχουν πεδία ή τομεί όπου δεν είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή ερμηνεία υπερτερεί για τα πρωτοβάθμια δικαστήρια. Μπορούν αυτά τα δικαστήρια να ξεκινήσουν μια προκαταρκτική διαδικασία και να ζητήσουν τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πώς ξέρετε ως νομική υπηρεσία ότι αυτό δεν θα είναι πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο επανειλημμένως έχει πει ότι υπάρχει αυτονομία ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαστικού συστήματος. Δεν το έχουμε θέσει το ερώτημα ρητά στο δικαστήριο, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Τώρα ο Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γιουρή, κυρία Γκέρινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάτι ακόμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας <clears throat> είναι και τα ζητήματα και οι συγκινήσεις οι οποίες δημιουργούνται στους πολίτες μας σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Οι πολίτες μας θα βγουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν πέραν της νομικής αυτής της γνωμοδότησης που έχουμε ακούσει και σε πείσμα αυτής της γνωμοδότησης ίσως υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για τα κοινά αυτά εργαλεία που έχουν να κάνουν με το ISDS. Αυτή τη στιγμή <clears throat> δεν έχουμε τη δυνατότητα να δεχτούμε την συμφωνία όταν υπάρχουν τόσο έντονες διαμαρτυρίες από τους πολίτες. Θα πρέπει να βρούμε μια απλή εξήγηση, εάν αυτό εφικτό, για το πώς <clears throat> το ISDS, το εργαλείο αυτό, δεν θα αποτελέσει μια απειλή για τους πολίτες μας, οι οποίοι φοβούνται αυτή τη συμφωνία και μια άλλη συμφωνία που είναι η TTIP και είναι και αυτή η υποδιαπραγμάτευση. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι, μήπως υπάρχει κάποια απλή εξήγηση η οποία καταδεικνύει ότι αυτή η συμφωνία συνάδει με τις ε, συνθήκες και δεν είναι απειλή για τους πολίτες. Η Μα... Μαρία Σάκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, <coughs> Πρόεδρε μάλλον, και σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που μας έχετε παράσχει. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περίπου 1.400 διμερείς συμφωνίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν εργαλεία όπως το ISDS. Έχει υπάρξει ποτέ προσβολή της ε, συμβατότητας αυτών των νομικών εργαλείων με τον ενωσιακό νόμο. Υπάρχει κάποια πρότυπη διαδικασία που ακολουθεί η Κομισιόν, που έχει ακολουθήσει η Κομισιόν, προτού προτείνει αυτή τη μορφή του ISDS. <clears throat> Θα ήθελα να πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι νομικές προτάσεις δεν γίνονται χωρίς να υπάρχει η αρμόδια βάση. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μάθουμε λίγο περισσότερο πώς έγινε η αξιολόγηση των προτάσεων της Κομισιόν και πώς οι νέες προτάσεις που αντανακλούν την πολιτική θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνδέονται με τις 1.400 συμφωνίες διμερούς χαρακτήρα για τις οποίες υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες ίσως και διαμαρτυρίες αλλά δεν έχει εγερθεί το θέμα της συμβατότητός τους με το κοινοτικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Ο κ. Uh, uh, uh, το, κύριο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη δική μου άποψη, είναι αν η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις διαμάχες και διαφωνίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή της Συμφωνίας ΣΥΤΑ και σε ποιο βαθμό οι αξίες και οι αρχές που περιλαμβάνονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να εξασφαλιστεί μετά από την θέση σε εφαρμογή της Συμφωνίας ΣΥΤΑ. Ευχαριστώ. Και τώρα η Αν Μαρή Μινέρ. Σας ευχαριστώ, λέει και η Αν Αυτό το οποίο με ανησυχεί για τη γνωμοδότηση αυτή είναι ότι δεν έχει αρκετό ειδικό βάρος. Γνωρίζουμε ότι γύρισε πίσω τρεις φορές μέχρι ότου να υπάρχει γενική ικανοποίηση για αυτήν την, ε, α, συμφωνία, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Αυτό το περιμένει κανείς από μια εταιρεία συμβούλων, αλλά όχι από ένα ανεξάρτητο νομικό σώμα. Δεν ξέρω γιατί όλοι είσαστε τόσο ικανοποιημένοι με την αντιμετώπιση αυτή για το ISDS. Ουσιαστικά μιλάμε για τη δημιουργία ενός νέου δικαστηρίου, ενός νέου νομικού συστήματος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το τωρινό ένομο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί κανείς να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Ένωση Δικαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναρωτιέται κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα, έχει την δικαιοδοσία καλύτερα να δημιουργήσει ένα τέτοιο νέο δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών δεν βλέπει να, υπάρξει, να υπάρχει ανάγκη για ένα περαιτέρω δικαστήριο, γιατί τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται εκεί έρχονται σε σύγκρουση <clears throat> με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Γερμανική Ένωση Δικαστών έχει εκφράσει την άποψή τη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενό νέου δικαστήριου. Θεωρεί ότι αυτό είναι ο λαθασμένο τρόπο για να εγγυηθούμε για τα δικαιώματα των δύο πλευρών. Και επίση, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να εισαγάγει το σύστημα ISDS, διότι περιορίζει τα δικαιώματα των κρατών μελών και των ενωσιακών νόμων και ένα περαιτέρω επιχείρημα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για το κατά πόσο η νομική τάξη της Ευρώπης θα πρέπει να υπόκειται στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί λοιπόν να υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα το οποίο θα δημιουργηθεί εδώ πέρα χωριστά από τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και έχουμε δει και την ερμηνευτική δήλωση για τη ΣΕΤΑ η οποία παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Δεν ξέρουμε <clears throat> ποιο είναι το καθεστώς αυτής της δήλωσης ε, στην ε, σύμβαση της ε, Βιέννης. Αλλά εγώ δεν είχα καμία ευκαιρία να λάβω το λόγο και να ρωτήσω σε σχέση με αυτή την ερμηνευτική διαδικασία. Κύριε Ροζιέ, είσαστε στον κατάλογο και έχετε ζητήσει το λόγο. Δεν μου είπαν ότι θα πάρω το λόγο. Ευχαριστώ πάντως. Συμφωνώ με τις επιφυλάξεις οι οποίες ακούστηκαν. Έχουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για τη συμβατότητα των διαιτητικών αυτών μηχανισμών. όπως έλεγε και η Κίρτον Ντάρτινγκ, έχουμε προηγούμενα σε επίπεδο νομολογίας και γι' αυτό έχουμε διαφορετική άποψη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διαρωτώ με πώς είναι δυνατόν να ξεκινήσει κανείς στην εφαρμογή ε, μιας τόσο περίπλοκης και αμφισβητήσιμης ε, ερμηνείας χωρίς να μιλήσουμε για το θέμα της ισότητας των ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και χωρίς να ζητήσει τη γνώμη ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εγώ δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Αυτή στιγμή ε, υπάρχουν αμφιβολίες γύρω από αυτό, ε, θα έπρεπε σίγουρα να ζητηθεί η γνώμη του δικαστηρίου. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Και εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για τη συμβατότητα της ρύθμισης που προτείνεται. Πρώτον, γιατί το, Ευρωπαϊκό, το δικαστήριο το ειδικό αυτό παραβιάζει την μονοπωλιακή αν θέλετε ή την αποκλειστική δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να κάνει την πρώτη ερμηνεία του πρωτογενούς δικαίου. Και δεύτερον, επίσης πριν φτάσουμε ακόμα σε αυτό το στάδιο, αγνοεί πολλές φορές τις πιθανές νομικές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, το θέμα έχει τεθεί ήδη από, το ίδιο, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 για τις διμερείς διαφορές και συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, λέγοντας ότι αυτού του είδους τα δικαστήρια δεν σέβονται το κοινοτικό δίκαιο και στην περίπτωση αμφιβολίας για την ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου δεν παραπέμπουν το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συνεπώς λοιπόν δεν έχουμε εγγυήσει ότι το διατητικό αυτό δικαστήριο ε, θα σεβαστεί το κοινοτικό δίκαιο. Τα επιχειρήματα λοιπόν δεν με πείθουν και καλύπτεται από τις ε, ρυθμίσεις και ένα μικρό τμήμα του κοινοτικού δικαίου. Τίθεται και θέμα λοιπόν στρέβλωσης και της ενιαίας αγοράς Νομίζω ότι κάποια συγκεκριμένα άρθρα της Συμφωνίας ΣΕΤΑ παραβιάζουν το 45, 49, 50 και 66. 56 συγγνώμη, της συνθήκης, τα οποία κινδυνεύουν να παραβιαστούν συστηματικά. Σαν παράδειγμα, μια γερμανική εταιρεία καναδικής ιδιοκτησίας στην ε, Γερμανία δεν μπορεί να μάλλον να προσφύγει σε νομική προστασία εθνική ενώ μια γαλλική επιχείρηση η οποία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά δεν έχει την δυνατότητα αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο και να μην υπάρχουν στρεβλώσεις εις βάρος των Ευρωπαίων εταίρων. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο κύριος Μαρίνο Πίντο, γιατί θέλουμε να φύγουμε από τη δημόσια δικαιοσύνη των δικαστηρίων, των δημόσιων δικαστηρίων. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να επιλύσει θέματα διαφωνιών σε ό,τι αφορά το δίκαιο των συμβάσεων. Υπάρχει αυτή της ε, δικαιοσύνης η οποία είναι παμπάλαια και οικουμενική και λέει ότι το δίκαιο το οποίο είναι εφαρμόσιμο είναι το δίκαιο του, της χώρας όπου γίνεται, όπου υπάρχει διαφορά. Υπάρχουν, χώρες, υπάρχουν λοιπόν αυτοί που θέλουν να κάνουν επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θέλουν να είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δικάσουν διαφορές. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η περιφρόνηση προς τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους δικαστές της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα διαιτητικά δικαστήρια υπάρχουν για να επιλύσουν διαδικασίες όταν υπάρχει μια, υπάρχει μια παρουσία αυτού του επίμαχου αδικημένου σε κάποια χώρα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί λοιπόν να υπάρξει πρόσβαση στα διαιτητικά δικαστήρια. Γιατί θεωρούνται ότι καλύτερα τα διαιτητικά δικαστήρια. Τι είναι αυτό που δεν μπορούν να κάνουν τα δημόσια δικαστήρια. Γιατί δεν μπορούν οι ανεξάρτητοι δικαστές στα κανονικά δικαστήρια να λειτουργήσουν. Ενδεχομένως μετά από μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο γρήγορα. Αυτά κάνει λοιπόν ένας, ένας ε, δικαστής είναι ανεξάρτητος, ενώ αυτοί οι οποίοι είναι οι διαιτητές σε αυτά τα δικαστήρια μπορεί να έχουν συνδέσει με τη μία ή με την άλλη επιχείρηση. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο και η ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου θα υπερέχει έναντι άλλων νομικών συστημάτων. Αν αυτά τα διαιτητικά δικαστήρια δεν υπόκειται στην δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πώ μπορούμε να ξέρουμε, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου και ομοιογένεια ερμηνεία. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απάντηση σε αυτή. Εμένα μου είπανε ότι δεν υπήρχαν περιορισμοί χρόνου για τα θέματα αυτά. Διαμαρτύρομαι. Όταν έχουμε μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να έχουμε το χρόνο για να μπορέσουμε να, να μιλήσουμε και να κάνουμε τι ερωτήσει, οι οποίε είναι απαραίτητε για να συζητήσουμε. Αν δεν θέλετε να έχουμε διάλογο, δεν έχει νόημα αυτό το οποίο κάνουμε. Χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Ναι, πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο. Καταλαβαίνω τα όρια του χρόνου, αλλά αυτό είναι και ένα τρόπο να εμποδίσουμε τη συζήτηση για ένα θέμα το οποίο είναι εξόχω σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι είπαμε ότι θα έχουν περιοριστεί σε δύο λεφτά. Πρέπει να ακολουθήσουμε. Με αυτό είναι λάθο, λέει ο κ. Μαρίνο Πίντα. Δεν είναι τρόπο συζήτηση αυτό. Δεν μπορούμε να συζητάμε και να μην συζητάμε στην πράξη, Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερις ερωτήσεις έχω να θέσω στην νομική υπηρεσία. Το γεγονός ότι προβλέπεται ότι πρέπει να εξαντληθούν τα εγχώρια ένδικα μέσα είναι τρόπος να ε, καθησυχαστούν οι αμφιβολίες που εκφράστηκαν προηγουμένως για το ISDS και το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων. Αυτό καταρχά. Κατά δεύτερον, δεν πρέπει να ρωτήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπάρχει συμβατότητα ή όχι. Η Επίτροπος Μάλστρομ και η σχετική Γενική Διεύθυνση λέει ότι αυτή η νομική οδός θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις νέες εμπορικές συμφωνίες. Από τη στιγμή που μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο δεν θα πρέπει το δικαστήριο να αποφανθεί και έτσι να ενισχυθεί αυτό το εργαλείο επίλυσης διαφορών επενδυτικών. Τρίτο ερώτημα. Εκτιμώ ιδιαίτερο στην αξιολόγηση της νομικής υπηρεσίας που λέει ότι ο οικονομικός αντίκτυπος δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη δυνατότητα του νομοθετήν του ρυθμίζει. Κοιτάξτε, τα κράτη-μέλη που έχουν τα μέσα να δώσουν αυτό τον οικονομικό αντίκτυπο μπορεί να μην έχουν πρόβλημα, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτές τις αποζημιώσεις, άρα ε, παρακολύονται εμφανέστατα στη δυνατότητά τους να νομοθετήσουν. Ή μήπω υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι να καλυφθούν οι επενδυτικοί κίνδυνοι. Γιατί τελικά περί αυτού πρόκειται, για τον επενδυτικό κίνδυνο. Π.χ. γιατί να μην έχουμε ασφάλειες να καλύψουν οι ασφαλιστικές τον επενδυτικό κίνδυνο, να καθησυχαστούν οι επενδυτές, να μην υπάρχει νομική ε, αβεβαιότητα. Είναι ένα ιδιωτικό σύστημα για τον ιδιωτικό τομέα και πληρώνει ο ιδιωτικό τομέα. Όταν είμαστε επιχειρηματίες παίρνουμε κινδύνους και μπορούμε να ασφαλιστούμε και για αυτού ε, Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί δεν έχει αξιολογηθεί αυτή η δυνατότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Εάν ένα, πάνω σε ένα πράγμα συμφωνούμε όλοι εμείς για το δικαστήριο είναι για το ότι δεν μπορεί κανείς να είναι απολύτως βέβαιος. Μπορεί να νομίζει ότι έχει μία υπόθεση ε, πανίσχυρη και σίγουρα θα την κερδίσει και μπορεί τελικά το δικαστήριο να αποφασίσει διαφορετικά. Σκέφτεται με το δικό του τρόπο. Εγώ Περιμένω με αγωνία την απόφαση του δικαστηρίου για τη συνθήκη του Μαρακές. Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστά τα επιχειρήματά μας, αλλά ποτέ κανείς δεν είναι σίγουρος. Τώρα, ως προς τη ΣΕΤΑ, τη και την προστασία των επενδυτών, είναι πολύ σοβαρές οι αμφιβολίες θεωρείται πολύ ότι δεν συνάδει με τις συνθήκες. Αύριο θα παρουσιαστεί μια δήλωση που υπογράφουν 100 Ευρωπαίοι καθηγητές νομικής και ο καθηγητής Κονσκινιμιέντη του Ελσίνκη και θα ενθαρρύνει η δήλωση αυτή τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο να αποκτήσουν τη γνώμη, να ζητήσουν τη γνώμη του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το κατά πόσο η ΣΥΤΑ είναι συμβατή με τις συνθήκες. Είναι πολύ καλύτερο να πάμε λοιπόν στο δικαστήριο πριν κυρώσουμε τη συνθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις προς την νομική μας υπηρεσία και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να απαντήσει. Η δική μας νομική υπηρεσία έκανε την ακόλουθη εκτίμηση. Είπε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διεθνείς συμβάσεις, έχει και την δυνατότητα να υπόκειται εφόσον το επιθυμεί σε διεθνή δικαστικά σώματα, τα οποία εννοείται ή προϋπήρχαν ή δημιουργούνται επί τούτου και τα συμβαλόμενα μέρη ε, δέχονται να υπόκειται στη δικαιοδοσία τους. Τώρα, το ερώτημα για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Ποιο είναι το Διεθνές Δικαστήριο το οποίο κανονικά θα είχε την δυνατότητα να ασχοληθεί με πιθανές συγκρούσεις ανάμεσα στους συμβαλωμένους. Genus Proximum, ένα αντίστοιχο συγγενές σύστημα στο οποίο θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε για να καταλάβουμε. Το Διεθνές Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος, οπότε δεν, είναι, δεν μπορεί να είναι αρμόδιο θα μπορούσαμε να γίνουμε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου. Εν ποιο είναι το γένος πρόξιμουμ στο οποίο υποκείμεθα. Αυτό ίσως να μπορέσει να διαφωτίσει τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Και δεύτερη ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ορισμένες δια... διαδικασίες επί παραβάση για παραβίαση ε, καθεστώτων ΦΠΑ στο εσωτερικό. Μήπως να υπάρχει κάποιο επίπεδο ομοιότητας με την περίπτωση που μας ενδιαφέρει, ίσως όχι, αλλά καλό θα είναι τέτοιου είδους αντίστοιχα διαιτητικά σώματα να δούμε τι, με ποιο τρόπο λειτουργούν σε ενδοκινοτικό επίπεδο. Ο κ. Λεμπετών. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή, η συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά προφανώς εμπεριέχει πολιτικά θέματα τα οποία θέλω να αναφέρω εδώ γιατί δημιουργεί μια αχαλήνωτη συμφωνία ε, ελευθέρων συναλλαγών που οδηγεί σε πολλά προβλήματα οικονομικά, φύγει το σύστημα ονομαζίας προέλευσης και οδηγεί σε πολλές ζημίες στη Γαλλική Γεωργία. Αλλά περνάω στο νομικά θέματα τώρα, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. ήταν λίγο πιστική, πολύ λίγο πιστική αυτή η νομική γνωμοδότηση και υπάρχουν τρία προβλήματα τα οποία παραμένουν. Το πρώτο πρόβλημα είναι φυσικά η ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου που φυσιολογικά είναι αποκλειστική δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και εδώ πέρα αυτή <clears throat> αποθείται γιατί το δικαστήριο που προτείνει σε τα θα πάρει αδίδυτα μία απόφαση και μία θέση για το ενωσιακό δικαίωμα χωρίς να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία προδικαστικής ερώτησης. Επομένως δημιουργείται ανταγωνισμός προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φυσικά μας είπαν ότι δεν θα υπάρχει κάποιο προηγούμενο, αλλά παρόλα αυτά πλήττει τις συνθήκες, παραβιάζει συνθήκες. Δεύτερο πρόβλημα είναι το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σαφές πρόβλημα <clears throat> διάκρισης προς όφελο των ξένων επενδυτών. Τι θα συμβεί. Αν συγκρίνετε την κατάσταση ενός ξένου επενδυτή με ένα Ευρωπαίο επενδυτή, σε περίπτωση ε, διαμάχης ο ένας θα έχει την πρόσβαση σε ένα χωριστό ειδικό δικαστήριο, ενώ ο Ευρωπαίος επενδυτής δεν θα έχει την ίδια δυνατότητα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα λοιπόν διακρίσεων και αναρωτιέται κανείς αν αυτό παραβιάζει ή όχι τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το τρίτο πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα κυριαρχικότητα των κρατών μελών. Κατά τη δική μου άποψη, η ΣΕΤΑ είναι μια μεικτή συμφωνία η οποία πρέπει να εγκριθεί και από τα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό δεν πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα, πρέπει να επιληφθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας κοιτάζει και σας βλέπει με αυτά που κάνετε η κοινή γνώμη. Μην κάνετε την Ευρώπη Ευρώπη των επιχειρηματιών και μόνο. Ο κύριος Σόλτς, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από τους συναδέλφους, αλλά θέλω να θέσω δύο ερωτήματα τα οποία φαίνονται από αυτά που είπε η νομική υπηρεσία, το πρόσθετο δικαστήριο θα αφορά μονάχα τα θέματα τα οποία προκύπτουν από την συνθήκη ΣΕΤΑ. Αλλά υπάρχει μια οριζόντια σύνθεση αυτή η σύνδεση αυτής της συμφωνίας με άλλες συνθήκες. Πώς λοιπόν θα ακολουθήσουμε αν παραγματικά η Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποιήσει το άρθρο 50 και δημιουργήσει μια χωριστή συμφωνία με τον Καναδά που θα είναι που θα έχει, αν κάνει ένα, μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει παρόμοιο χαρακτήρα, πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αν υπάρξει μια αντίστοιχη συμφωνία με την ε, Μεγάλη Βρετανία. Αυτό φυσικά ενδιαφέρει και τους ξένους επενδυτές αλλά ενδιαφέρει και τους ε, Ευρωπαίους ε, επενδυτές. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να, εξασφαλιστεί, να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτών των επενδυτών έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των κρατικών ε, επιδοτήσεων που παρουσιάζονται ως πρόβλημα. Δηλαδή, όταν στη δήλωση για την Συμφωνία ΣΕΤΑ που θα εγκρίνει το Συμβούλιο για να δημιουργήσει νομικά αποτελέσματα, τίθεται το θέμα για τις δημόσιες ε, προμήθειες, για τα πρότυπα σε οικολογικό κοινωνικό επίπεδο. Κατά πόσο λοιπόν αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσβολής από ξένους επενδυτές και πώς αυτό θα σημάνει ότι υπάρχει ίση αντιμετώπιση των ξένων επενδυτών και των επενδυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτό συνάδει με την έννοια της κυριαρχικότητας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ προσεκτικός γιατί η νομική υπηρεσία είναι ακριβώς πίσω μου και θα προσπαθήσω να μην την προσβάλλω. Δεν θα είμαι πονηρός, αλλά θα πω ότι όταν τελικά ε, κανείς αναγκάζεται να το αφαιρέσει το λόγο μετά από 10 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι το θέμα είναι πολύ πιο περιπλοκό από ό,τι φαίνεται ή από ό,τι νομίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ε, δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι οι νομικές πτυχές. Η νομική ασφάλεια και ο αγώνας ε, ενάντια στις αβεβαιότητες είναι ο ακρογωνιαίος λήθος ενός κράτους δικαίου. Και το ερώτημα που θέτω στο Κοινοβούλιο και που δεν θέτω στη νομική υπηρεσία, γιατί είναι πολιτική απόφαση, είναι το εξής γιατί φοβόμαστε και τι φοβόμαστε και δεν προσφεύγουμε στο δικαστήριο για να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Αφού όλοι συμφωνούμε και λέμε ότι υπάρχει νομική δυσκολία, υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών, ας παραμείνουμε στην πολιτική ε, θέση λοιπόν του ναι ή όχι είναι καλό πράγμα η ΣΥΤΑ, και εντωμεταξύ ας προσφύγουμε στο όργανο που μπορεί να αποφανθεί και μπορεί να διαλύσει τις νομικές αμφιβολίες, τις οποίες δεν θέλουν ούτε οι επενδυτές. Ας κριθεί λοιπόν αυτό το θέμα δικαστικά, κατά πόσο υπάρχει συμβατότητα, από το δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κασπάρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, το άρθρο 7 στην Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπάρχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Αν εμείς δεν εφαρμόζουμε αυτό το άρθρο δεν έχει κανένα νόημα η Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όλοι συμφωνούν ότι στις διεθνείς μας συμφωνίες δεν θα πρέπει να παραβιαστεί το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Αλλά η δυνατότητα να έχουμε, διδα, ε, <clears throat> να έχουμε δικαστήρια, δεν τα δεχόμαστε. Αλλά δεν δεχόμαστε να αλλάξουμε το, ε, το, το νομικό μας σύστημα. Επομένως, στην πράξη δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση και επομένως θα πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεύτερον, εγώ εντυπωσιάζομαι πολύ, έχουν εκφράσει μια άποψη η οποία είναι αρνητική. Αυτοί οι οποίοι έχουν αρνητική άποψη θα έπρεπε να είχαν απορρίψει όλες τις ε, συμφωνίες του παρελθόντος που αυτοί λοιπόν που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία δεν ήθελαν και καμιά προηγούμενη συμφωνία ακόμα και αν δεν είχε διαδικασία για την επίλυση των διαφορών μεταξύ ε, επενδυτών και κρατών. Και οι 1.400 συμφωνίες που έχουν συναυθεί σε διμερές επίπεδο έχουν καταδείξει ότι λειτουργεί πολύ καλά αυτό το εργαλείο, μόνο σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν αμφίβολες αποφάσεις. Έχουν καταδείξει λοιπόν οι 1.400 συμφωνίες ότι δεν υπήρξε πρόβλημα να μη συνάδει η απόφαση ενός δικαστηρίου με το εθνικό δίκαιο και δεν υπάρχει καμία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι είναι προβληματικές αυτές οι αποφάσεις των διαιτητικών δικαστηρίων και αυτή η βάση λοιπόν που αναφέρει η νομική υπηρεσία μας είναι πολύ ορθή και επομένως δεν πρέπει να περιορίσουμε τη δυνατότητα διαιτητικού δικαστηρίου και σας παρακαλώ να σταματήσετε αυτά τα επιχειρήματα που λέτε σε σχέση με το δικαστήριο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει Ξαναγυρίζουμε προ την Κομισιόν. Κύριο Μπάουμ έχει το λόγο. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκια. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά το πώς εφαρμόζεται η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ήδη εξ αρχής από το 2010 αρχίσαμε να εξετάζουμε τα θέματα αυτά το σύστημα το οποίο έχουμε μπροστά μας διαφέρει από την Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό είναι και ζητούμενο. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω πέντε σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη. Έχουμε να κάνουμε με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχει σε διεθνείς συμβάσεις με συγκεκριμένα μέσα επίλυσης διαφορών. Αυτό ισχύει και για τον Καναδά και για όλες τις χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμεθα. Κίνα, Ινδία και τις υπόλοιπες χώρες. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η νομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι ταυτόσημη και έρχομαι εδώ και σε κάποιες από τις ερωτήσεις με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούμε για όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Δηλαδή ένα σώμα αναγνωρισμένο από τον ΠΟΕ και αντίστοιχα σώματα σε όλες τις ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το δικαστήριο εξετάζει με βάση το κοινοτικό δίκαιο σαν γεγονός. Δεν τίθεται θέμα ερμηνείας του κοινοτικού δικαίου, αλλά η συμφωνία στα πλαίσια των ΠΟΕ εξετάζει με βάση τις ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου και αυτό δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα συμβατότητας. Το σύστημα λοιπόν της ΣΕΤΑ και το σύστημα σε όλες τις συμφωνίες οι οποίες διαπραγματεύτηκαν στο, έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευση στο παρελθόν εξετάζεται το κοινοτικό δίκαιο σαν γεγονός όχι από μεμονωμένα κοινοτικά όργανα και δεν δίδονται ερμηνείες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αντίθετες ή δεσμευτικές για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς ε, δεν είναι ρόλος μας να εξηγήσουμε ακριβώς, αν και το έχουμε κάνει γραπτά, γιατί οι Γερμανοί νομομαθείς και η άλλη ομάδα των Ευρωπαίων νομομαθών εδώ κάνουν ένα λάθος. Ε, σε σχέση τώρα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς η θέση σε σχέση με τα ανώτατα δικαστήρια των υπόλοιπων συμβαλωμένων χωρών. Το ανώτατο δικαστήριο του Καναδά, το ανώτατο δικαστήριο της Κίνας θεωρούν ότι έχουν αρμοδιότητα και μονοπόλιο για την ερμηνεία του δικού τους εθνικού δικαίου και δεν συμμετέχουν, ε, δεν αμφισβητούν την συμφωνία ε, γιατί το σύστημα ISDS δεν οδηγεί σε δεσμευτικές ερμηνείες εθνικού δικαίου. Το τέταρτο σημείο τέθηκε από δύο από τους συναδέλφους σας είναι το θέμα των διακρίσεων. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι οι επιχειρήσεις που μπορούν να ανακινήσουν τέτοιες επιχειρήσεις στην Ένωση το κάνουν επειδή είναι καναδικές. Μπορούν να το κάνουν επειδή είναι καναδικές, είναι καναδικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορούν να το κάνουν αν ήταν γαλλικές ή αγγλικές. Και αυτό γιατί ε, αντίστοιχα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τα ίδια δικαιώματα στον Καναδά και μπορούν να προσφύγουν στον Καναδά. Και το ίδιο ισχύει και με τις άλλες διεθνείς συμφωνίες. Τίθεται λοιπόν θέμα αμοιβαιότητας και η αμοιβαιότητα είναι συστατικό θεμέλιο γενικά όλων των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων. Και οι περιορισμοί που μπορεί να τίθενται, τίθενται σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου μόνο αν υπάρχει λόγος αμοιβαιότητας. Τώρα για το αν μια ευρωπαϊκή επιχείρηση δημιουργήσει μια επιχείρηση στον Καναδά για να διεκδικήσει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τέτοια παραθυράκια. Τώρα, η ύπαρξη των διατηρητικών σωμάτων και η συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση για τέτοιου είδους BIT στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι δύο τα διαφορετικές καταστάσεις σε σχέση με, τις, ε, με τα σώματα αυτά στο εσωτερικό των χωρών της Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ΣΕΤΑ λοιπόν και οι άλλες συμφωνίες μας παρέχουν πλήρη ελευθερία σε σχέση με τις διακανονιστικές ρυθμίσεις και είναι απόλυτα συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Λοιπόν, τώρα θα δώσω το λόγο, όχι πάνω από πέντε λεπτά, στην νομική υπηρεσία, να δώσει απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα περισσότερα από τα νομικά θέματα τα οποία γέλσαν έχουν αντιμετωπιστεί από τη νομική γνωμοδόση και από την προφορική μου παρουσίαση. Δεν πρόκειται ένα διαιτητικό δικαστήριο να ερμηνεύσει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εξήγησε και η Κομισιόν. Και πράγματι, τέτοιο θέμα δεν υπάρχει ήδη υπάρχουσα ε, ερμηνεία του κοινωνικού δικαίου. Δεν υπάρχει σύστημα προδικαστικής ερώτησης γιατί δεν μπορεί το δικαστήριο να ερμηνεύσει το ευρωπαϊκό δίκαιο παρά μόνο ως δεδομένο. Τι γίνεται τώρα αν υπάρχει κάποια προσβολή προς τη ΣΕΤΑ και φανεί ότι είναι παράνομη. Τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα βάσει του νόμου των επενδύσεων για να σταματήσει η ισχύ αυτή τη συμφωνία και να υπάρχει επαναδιαπραγμάτευση. Και επίση υπήρξε ένα ερώτημα ότι υπάρχουν αυτές οι 1.400 συμφωνίες, αυτό ήταν αντικείμενο σχολείων και από την Κομισιόν, έχουμε ένα σύστημα λοιπόν το οποίο υπάρχει ήδη, δεν είναι καινούριο σύστημα, το σύστημα ISDS το οποίο θα δημιουργηθεί εκ του μηδενός, πρέπει να το δούμε στο, στο πλαίσιο των ήδη υπαρχουσών συμφωνιών. Κάποιοι ομιλητέ αναφέρθηκαν επίση στην ανάγκη να θέσουμε ένα ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν βρίσκεται μέσα στη, νομική μας ε, ε, άποψη, γιατί δεν μας ρώτησε κανένα για αυτό το θέμα. Δεν υπησέρχομαι λοιπόν για αυτό το ζήτημα. Δεν μπορώ να παραθέσει σε αυτό. υπήρξε και ένα θέμα για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου γενικά. Λογικά αυτές οι συμφωνίες έχουν δυνατότητα επίλυση διαφορών μέσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Και οι διμερείς συμφωνίες, αυτό το θέμα το έθιξε η Κομισιόν ήδη, οι διμερείς συμφωνίες επενδύσεων, BIT, και με αυτά και με την αναφορά προς την ε, νομική μας γνωμοδότηση που είναι δημόσια, βρίσκεται στο διαδίκτυο. Μπορώ να κλείσω. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι να σας βοηθήσουμε αν χρειάζεται. Ε, Ευχαριστώ πολύ την νομική υπηρεσία. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Γιούρη για την ε, παρουσία της εδώ. Νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Είναι πάρα πολλές οι αβεβαιότητες. Θα παραμείνουμε σε επαφή. Ίσως έχουμε και διμερή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ, Σβόμποντα. Ο Σβόμποντα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κοινή ακρόαση της νομικής υπηρεσίας. Να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής Γιούρη ότι εμείς θα πάμε, ότι θα πάμε στην αίθουσα ASP 3E2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ίντα. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά διάλειμμα και μετά θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία.